So, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten heute pünktlich, weil wir nämlich... Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε βέβαια πολύ άριθμοι εδώ σήμερα και έχουμε και πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό ας ξεκινήσουμε καλύτερα στην ώρα μας. Και αρχίζουμε αμέσως με το σημείο αριθμός 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 7 έχει αναβληθεί που πρόκειται για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Και Η ψηφοφορία για το σημείο 17 αναβάλλεται επίσης. Η έκθεση δηλαδή Κάντενβαχ. Στη συνέχεια έχουμε την έκθεση Σνέλχαρτ. Έχουμε προβλέψει... Α, δεν υπάρχει διερμηνία στα Ιταλικά, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει διερμηνία τώρα. Ρωτάει ο Πρόεδρος. Εντάξει, κύριε Γιαμπόρσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα σήμερα να σας παρουσιάσω την κατάσταση όσον αφορά εμένα τουλάχιστον για την έκθεση αυτή. Να ξέρετε ότι έχω εκπλαγεί και όσο καιρό ήμουν εδώ στο Κοινοβούλιο ποτέ δεν βρέθηκα αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω περί τίνος πρόκειται. Η DNA, μια, μια κυβερνητική οργάνωση η οποία χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση σε συνεργασία με σκιώδη εισηγητή από τους σοσιαλιστές με κατηγόρησε ότι δουλεύω για τα συμφέροντα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εσείς όλοι όσοι έχετε συνεργαστεί με τέτοιες εκθέσεις ξέρετε ότι έχουμε πάρει προτάσεις, έχουμε πάρει από τους λόμπις, από τις ομάδες πίεσης, διάφορες ιδέες από μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης. Κάπου 220 προτάσεις έχω ακούσει και υπάρχει και ο πίνακας του κυρίου Μάτσας Χάρτον, ο οποίος δουλεύει για την ε, οργάνωση την Ευρωπαϊκή για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά βασίζομαι επίσης και στα Ηνωμένα Έθνη και τις δικές τους διατάξεις όσον αφορά την ηχορύπανση. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποίησα όλα αυτά τα στοιχεία και χρησιμοποίησα τα νούμερα εκείνα τα οποία, στα οποία καταλήξαμε σε συμβιβασμό μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιομηχανίας και πολιτικών ομάδων. Τώρα λοιπόν αντιτίθεμε σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί σε βάρος μου και σε βάρος της δουλειάς μου. Εγώ χρησιμοποίησα τέσσερις ίδιους πίνακες. Ο ένα είχε τι αρχικέ προτάσει του Κέχαρτη, άλλη είναι της συναδέλφου Μέρκης. ο τρίτος πίνακας είναι ο δικό μου συμβιβασμό και ο τέταρτος πίνακας έχει να κάνει με τα ίδια δεδομένα περίπου, όπως και τα δεδομένα της κυρίας Μέρκης. Η κατάσταση έχει ήδη προχωρήσει πολύ και γι' αυτό ήθελα να ενημερώσω τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για αυτή την υπόθεση και να απευθυνθώ και στους κοσμήτορες. Μια που πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην κορυφή μιας ε, εκστρατείας της φήμησης του ατόμου μου. Πιστεύω ότι κάποιος έχει μάλιστα παρέμβει και στο site της ε, Porsche ε, παράνομα. Εκεί αναφέρεται το δικό μου βιογραφικό, αναφέρονται εκεί και διάφορα στοιχεία, οικονομικά και άλλα. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια εκστρατεία λοιπόν η οποία θέλει να δείξει ότι εμένα με πληρώνει η Πόρσε. Μια τέτοια συμπεριφορά λοιπόν ξεπερνάει τα όρια νομίζω του θεμητού ανταγωνισμού και ξεπερνάει και οτιδήποτε έχω συναντήσει στην καριέρα μου μέχρι σήμερα και γι' αυτό αποφάσισα να προσφύγω κατά γνώστων για την υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Έχουμε αναβάλει την έκθεση από την ημερήσια διάταξη και οι περιστάσεις που εξηγήσατε μόλις θα διερευνηθούν και μετά θα συνεχιστεί η εργασία επί της εκθέσεως. Τώρα, εγώ σας διάβασα πριν λίγες αναβολές. Το απόγευμα θα έχουμε το 4. Μετά την έκθεση Γκαρντίνη, Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Μετά θα κάνουμε την ψηφοφορία μας από 10 και 30, 12 και 30. Ο πρόεδρος δεν έχει μικρόφωνο δυστυχώς. Μετά Σόνικ, Κάμπαχ, Γιόργενσεν, Ματίας και Χάουκ. Αυτά για το πρωινό. Το απόγευμα συνεχίζουμε στις 3 μέχρι τις 5 προβλέπονται ψηφοφορίες. Horizon 2020 και πάλι ξανά Horizon 2020, μετά οι εκθέσεις και μετά το 28 η υπόθεση της μεθανόλης στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτά για την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και προχωρούμε Έχουμε βέβαια τους διερμηνείς, όπως γνωρίζετε, στις διάφορες γλώσσες και τα ελληνικά βεβαίω όπως ακούτε και μια ομάδα επισκεπτών που ακόμα δεν έχει προσέλθει από το Ροσκίλντε προσκεκλημένη μιας Γερμανίδας βουλευτού και για την έκθεση Sonic για το shale gas θα είναι παρούσα και μια ομάδα λήψεων τηλεοπτικών εικόνων και για το τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης θα έχουμε τσεχική τηλεόραση παρούσα εδώ. Τώρα υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις, ε, αλλαγές μάλλον σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους. Ο κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους από την Κύπρο. θα αντικαταστήσει τον κύριο Μαυρονικόλα ως αναπληρωματικό μέλος. Και σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τώρα τα πρακτικά της 20ης και 21ης έκτου και της 9ης 17ης εβδόμου είναι διαθέσιμα επιγραμμικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ψάχνετε να τα βρείτε σε έγγραφη μορφή ε, έξω από την πόρτα. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι το ψήφισμα για την 18η διάσκεψη του Κατάρ Κάνουμε τη σχετική προπαρασκευαστική συζήτηση για το πώς θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιε θα πρέπει να είναι οι θέσεις μας για τη μελλοντική πολιτική του κλίματος. Χαίρομαι γιατί έχει γίνει ευρύ το ψήφισμα είναι ένα είδος reality check και αμφισβητεί και την πολιτική μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα πρέπει να κάνει και η Κομισιόν, και ανοιγόμαστε περισσότερο και διεθνώς. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια διπλωματία του κλίματος. Έχω έρθει σε επαφή κατ' επανάληψη με την τώρα διαμορφούμενη υπηρεσία εξωτερικών δράσεων που νομίζω ότι θα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Δεν είναι μονάχα θέμα δηλαδή ενός ή δυο θεσμικών οργάνων, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί, όπως είπα, μια κλιματική διπλωματία και από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν και τεράστια κενά ανάμεσα στις θεωρητικές τιμές που ακόμα ελπίζουμε να επιτύχουμε και στην πραγματικότητα. Τα κενά αυτά, η απόσταση αυτή πρέπει να μειωθεί, διότι όλη αυτή η υπόθεση της αλλαγής του κλίματος έχει ένα κοινό στοιχείο. Το, για να αλλάξει το κλίμα ή να ανασταλεί αυτή η αλλαγή του κλίματος χρειάζεται χρόνος, πολύ, πάρα πολύ. Επειδή γνωρίζουμε την κατάσταση, μιλούμε για αντιδράσεις από πλευρά κλίματος σε χρόνο της τάξης των 20-25 ετών. Και αυτό Ε, γιατί, και αυτό γιατί αγνοούμε τις επιταγές της επιστήμης, οι οποίες έρχεται και μας λέει τι πρέπει να γίνει και εμείς, όπως είπα, σε παγκόσμιο επίπεδο τις αγνοούμε. Στο ψήφισμα αυτό, στο σχέδιο ψηφίσματος, έχουμε περιλάβει και τις αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες. Για τις εναέριες υπάρχει νομοθεσία. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο υπήρξε τότε ιδιαίτερα θαραλέο και περιέλαβε και την διεθνή διάσταση αυτού του φορέα μεταφορών. Τώρα αυξάνει η πίεση έτσι ώστε και οι διεθνείς οργανώσεις όπως η ΚΑΟ αλλά και η ΑΕΜΟ για τα πλοία, για τις θαλάσσιες μεταφορές, έχει αρχίσει η συζήτηση και προχωρεί, ώστε να, έχουμε, να, αποκτήσουμε ένα διεθνές σύστημα γιατί μόνο με διεθνές σύστημα θα μπορέσουμε να μειώσουμε ριζικά τις εκπομπές καυσαέριων. Καλά είναι εμείς να δουλεύουμε εδώ στην Ευρώπη, αλλά το 2010 ήμασταν εμείς υπεύθυνοι για 11% παγκοσμίω των αερίων του θερμοκηπίου, εμείς οι Ευρωπαίοι. Το υπόλοιπο 89% παράγεται αλλού. Άρα λοιπόν μόνο η διεθνής διάσταση μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία. Το έγγραφο, δηλαδή την ε, έκθεση αυτή, την έχουν συνεπεξεργαστεί πολλοί συνάδελφοι. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον συνεισηγητή Καρλ Χάιντ Φλόρεντς. Εσείς κάνατε ήδη, κύριε Πρόεδρε, την εισαγωγή Δυστυχώς τώρα θα σας τα πω λίγο στα τυφλά, αν μπορώ να το πω έτσι, διότι έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου. Να δούμε πού θα καταλήξουμε, όπως είπα θα είναι πτήση στα τυφλά. Πάντως χαίρομαι που έχουμε φτάσει και συζητούμε ξανά το θέμα. Ε, μιλήσαμε για την πλατφόρμα Durban, η οποία μπορεί να μας ικανοποιεί ή και όχι, πάντως το γεγονός είναι ότι υπάρχει μια πλατφόρμα τώρα, όπου όλοι μπορούμε να βασιστούμε και βέβαια έχουν γίνει λίγα βήματα, σχετικά λίγα βήματα και εκφράζω τη λύπη μου και εγώ όπως το είπε άλλωστε και ο Πρόεδρος ότι συντάσσουμε ωραία εξαιρετικά έγγραφα αλλά λίστα με η, λίστα των πραγματικών πεπραγμένων των πραγματικών αποτελεσμάτων είναι πάρα πολύ σύντομη. Και είναι σημαντικό να σκεφτούμε και τι ζητούμε και βεβαίως αυτά που ζητούμε να τα ζητήσουμε με ένταση δεν ε, υπάρχει κανένα σχετικό θέμα αλλά πρέπει να μείνουμε και στα πλαίσια του ρεαλιστικού. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Βέβαια, ορισμένοι θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν. Αλλά να φτιάξουμε και μια λίστα για το τι πετύχαμε μετά από τα δύο ή τρία αυτά χρόνια. Για μένα αυτό είναι σημαντικό, ακόμα σημαντικότερο. και εγώ ανησυχώ ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι θα γίνει στο μέλλον. Το Κιώτο 2 είναι προσωρινή υπόθεση και ε, αναρωτιέται κανείς πότε θα τη Για τα συγκεκριμένα θέματα τώρα αρχίζω με τα CDM για παράδειγμα γνωρίζω ότι υπάρχει ε, ασκείται πολύ κριτική, αλλά θέλουμε όντω να τα αφήσουμε να λήξουν ιδίω οι χώρες εκείνες που ασκούν καινοτομία στον τομέα της προστασία του κλίματο προσφέρουν πολλά και εγώ θα θεωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα λυπηρό να εγκαταλείψουμε τον τομέα αυτόν. Νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί. Το δεύτερο είναι ότι με τα λεγόμενα AAUS, με τις ποσοστώσεις δηλαδή για το διοξίδιο του άνθρακος, έχουμε σημαντικά πλεονάσματα στην Ευρώπη και πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτά ήταν θέμα διαφωνίας και μέσα στην Ένωση. Τότε υπό Πολωνική Προεδρία ο Προεδρεύων, ο Πολωνός Προεδρεύων είχε φανεί αρκετά άκαμπτος. Πρέπει ωστόσο να τα πούμε καθαρά τα πράγματα αυτά, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να τα δεχθούμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να υπερβούμε τα εσκαμένα, αν μπορώ να το πω έτσι, να έχουμε και νέα έκθεση IPECC Πρέπει να δώσουμε μια νέα πορεία στο όλο το τομέα αυτό. Ίσως να κάνω και λάθος. Η επιστήμη μας λέει ότι το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος γίνεται χειρότερο. Αλλά οι δραστηριότητες στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο νομίζω ότι έχουν μπει μια φάση πτώσης. Μακάρι να κάνω λάθος αλλά η καθημερινή ζωή μου δείχνει ότι έτσι είναι. Α, τώρα μου φέρνουν τα γυαλιά, τι ωραία. Ευτυχώς. Τι να κάνουμε, ανθρώπινες αδυναμίες. Πολύ ωραία, τώρα μπορώ καλύτερα να σας τα πω. Η πλατφόρμα λοιπόν που αναπτύξαμε στην τελευταία διάσκεψη πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να πούμε σαφέστερα τι γίνεται με τους χρηματοδότες. Είναι πραγματικά τόσο καλοί όσο υποστηρίζουν στα διάφορα έγγραφά τους. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Όχι μόνο χρήματα του δημοσίου. Πρέπει να αναζητηθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δεν είναι όμως μόνο τα λεφτά. Είναι και το λεγόμενο capacity building και η τεχνολογία που είναι πολύ σημαντικά. Η τεχνολογία βέβαια δεν είναι δωρεάν. Αυτό είναι σίγουρο. Και γι' αυτό τι, αυτό το προβάδισμα που διαθέτουμε πρέπει να το διατηρήσουμε στην τεχνολογία. Αλλά πρέπει να είναι δυνατό να γίνει και μεταφορά τεχνολογίας. Και να πωλείται, να μεταφέρεται και σε άλλες χώρες. Επίσης δεν με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διασκέψεις αυτές. Βέβαια ο, ο πρέπει να τα διορθώσει αυτά τα πράγματα. το να καθόμαστε σε μία αίθουσα με προσώπους 192 χωρών και να προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μία κοινή θέση, ε, δεν μπορεί αυτή παρά να είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό κοινό παρονομαστή. Το ίδιο ισχύει για την Ευρώπη. Για να πετύχετε ομοφωνία στο Συμβούλιο χρειάζεστε 27 ε, χώρες μέλη. Ένας μόνο, ένα, ένας μόνο τον ενοχλεί το στομάχι του εκείνη την ώρα και θα πει όχι και τελείωσε τότε η ομοφωνία. Πήγε περίπατο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πιο μακροπρόθεσμα θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας και ρεαλιστικά εργαλεία που να μπορούμε να δράσουμε με πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ πάντως τις και τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία ε, για το έγγραφο. Υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα στο κείμενο. Θα συμπληρώσουν βεβαίως οι διάφορες, οι διάφορες πολιτικές ομάδες και άλλα πράγματα. Πάντως Εν τέλει, έχω βάλει εγώ στο τέλος την γράφω δηλαδή μια λίστα που θα μπορούμε να πούμε σε δύο χρόνια ήδη ποια πράγματα έχουν επιτευχθεί και να βάλουμε το σχετικό σημαδάκι δίπλα. Αυτό ο κατάλογο ίσω είναι ωραίο, αλλά ούτε καν στην Ευρώπη δεν τον δέχονται πάντα. Τότε θα τον κάνω τον κατάλογο, προσπαθώ να τον κάνω τον κατάλογο πιο ρεαλιστικό. Αλλά αυτά που θα πρέπει, να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει εν τέλει να τα κάνουμε. Αυτό, από αυτό εξαρτάται πολύ και η, η αντίδραση των ε, πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα βλέπουμε όλοι καλύτερα μετά από τον τρόπο που μας τα εξηγήσατε. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον Καρλ Χάινς. Δυστυχώ έχετε δίκιο. Πιστεύω κι εγώ ότι από την επιστήμη γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Από την επιστήμη γνωρίζουμε ότι η πραγματικότητα είναι μάλλον χειρότερη από αυτό που φανταζόμασταν. Οπότε τα χειρότερα σενάρια ακόμα που είχαμε στη προηγούμενη έκθεση από το IPCC θα αποδειχθούν πολύ αισιόδοξα πράγματα. Επίσης είναι μάλλον δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό, ότι αυτά που πετύχαμε στην περσινή διάσκεψη, την 17, τελικά δεν μας βοήθησαν καθόλου. Κάποιοι είπαν ότι ήταν μεγάλη επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι καταφέραμε για πρώτη φορά να καταφέρουμε διάφορες χώρες να συνυπογράψουν σε μια δεσμευτική συμφωνία. Αν δούμε μεμονωμένα αυτό το ζήτημα, ναι, εντάξει, είναι θετικό βέβαια το ότι αναγνωρίζουν τώρα πως ε, έτσι πρέπει να είναι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κοιτάει μεμονωμένα αυτό το πράγμα, πρέπει να δει πότε θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Δυστυχώς λοιπόν η δεσμευτική συμφωνία, ο δεσμευτικός στόχος μιλάει για το 2015 το πολύ αλλά αυτό σε όρους ΟΙΕ σημαίνει το νωρίτερο στην ουσία. Λέει ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει παρά το 2020. Άρα το νωρίτερο το 2020 για μένα. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο για μένα ότι δεν φτάνουν όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να μειώσουμε το 2020 ανάμεσα σε 25 και 40% ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τότε έχουμε 50% πιθανότητες να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς που είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε καν πιθανότητες 50% να σταθεροποιήσουμε τη θερμοκρασία. Και δύο βαθμοί, λένε οι επιστήμονες, είναι μάλλον πολύ φιλόδοξο. Οπότε, ειλικρινά, υπάρχουν πολλοί λόγοι εδώ να πιέσουμε περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το ψήφισμά μας είναι ισορροπημένο, πιστεύω. Πιστεύω επίσης ότι επικεντρωνόμαστε σε πολλά καλά θετικά στοιχεία, κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και συμφωνώ και με τον Πρόεδρο που είπε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και με άλλους τρόπους να επηρεάσουμε την κατάσταση, με την περιβαλλοντική διπλωματία για παράδειγμα. Αλλά να σας πω και δύο λόγια που μπορεί να μην είναι πολιτικά ορθά, αλλά αυτό που έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση με την Πολωνική Προεδρία ήταν ένα σκάνδαλο. Τελικά εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της Πολωνίας και όχι της Ευρώπης. Αν ξανασυμβεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι πλήττεται η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα μπορούμε πια να μιλάμε με μία φωνή. Εννοείται. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Επίση, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά. Είναι κάτι που το συζητάμε βέβαια χρόνια και χρόνια. Πολλοί εδώ μέσα πίστεψαν ότι με τη νέα συνθήκη θα υπήρξε μια τέτοια συμφωνία και θα συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις. Ε, δεν έγινε αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μας σέβονται στο ελάχιστο τουλάχιστον, ώστε να συμπεριλάβουν εμάς ή έστω τον πρόεδρό μας τις συντονιστικές ε, συνεδριάσεις, έστω ως παρατηρητές. Θα ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί να μην μπορεί ο Πρόεδρός μας να βρίσκεται παρόν στις ε, συντονιστικές αυτές συνεδριάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Χάση είναι επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συμφωνώ και με τον Καρλ Φλόρενς και με τον ε, Γιώργενσεν για το μήνυμα των επιστημόνων. Και εγώ έχω συζητήσει με ειδικού για το κλίμα και αυτά που μου λένε είναι πολύ ανησυχητικά. Όσοι συνομιλητές είχα, είπαν ότι αυτό το, αυτός ο στόχος του 2% είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Στα περιθώρια να τον πετύχουμε είναι ελάχιστα δεδομένες της κατάστασης στη βιομηχανία. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να δράσουμε. Όλοι ακούσαμε τα φετινά νέα για την ε, Αρκτική, για τους πάγους που λιώνουν εκεί. Η διαφορά με πριν από πέντε χρόνια είναι τεράστια. Πριν από ε, πέντε χρόνια που είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ήδη ήταν το νέο στα μέσα ενημέρωσης. Φέτος που είχαμε μια νέα στιβάδα πάγων που έλειωσε πέρασε στα ψηλά. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε ισχυρό ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Όλα τα βήματα που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα έχουν αναλυθεί ακριβώς επειδή υπήρξε ευρωπαϊκή ηγεσία. Φέτος, στην ε, διάσκεψη, ίσως υπάρχουν και νέα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Μια επίσημη απόφαση για να ξεκινήσει η δεύτερη ε, περίοδος δέσμευσης μετά το Κιώτο. Και χρειάζεται κάποια απόφαση για τις ε, καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες, τα AAUs. Τι εμπόδιο υπάρχει και το Συμβούλιο. Έχει αυτή την παράδοση να υιοθετεί συμπεράσματα ομόφωνα. Δεν υπάρχει τέτοια βάση στις συνθήκες. Ακόμα και πριν την Λισαβόνα δεν υπήρχε τέτοια βάση. Γιατί να αποφασίζει ομόφωνα λοιπόν το Συμβούλιο για θέματα που έχουν να κάνουν με διεθνείς διαπραγματεύσεις. Μετά τη Λισαβόνα ακόμα λιγότερο λοιπόν. Πρόκειται απλώς για μια παράδοση, μια κακιά συνήθεια που έχουν. Έτσι θέλουν να πιστεύουν ότι τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν ομόφωνα. Είναι για μένα ξεκάθαρο πια ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και ισχυρή όσο θα θέλαμε αν δεν πάψει να ισχύει αυτός ο κανόνας εντό αγωγικών της ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Πρέπει να αποφασίζουν με δική πλειοψηφία. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Ένα από τα θέματα γενικά είναι να κλείσει το χάσμα των μεγατόνων, δηλαδή ανάμεσα στις εθνικές δεσμεύσεις και σε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς. Θέλω να ξέρω τι πρόοδος έχει επιτευχθεί για αυτό το θέμα, τι περιμένουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω συμμετάσχει σε τρεις διασκέψεις για το κλίμα. Και πάντοτε έχουν ένα έντονο δραματικό χαρακτήρα, δηλαδή οι προετοιμασίες είναι πάρα πολύ σκληρές και δύσκολες. Το ίδιο συμβαίνει και τούτη τη φορά. Είδαμε ότι στην προπαρασκευαστική διάσκεψη στην Βόνη ούτε επί της διαδικασίας δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και δεν προχωρήσαμε καν στην ουσία. Τώρα στην Μπανκόκ τα πράγματα πήγαν λίγο καλύτερα, αλλά πάλι ο χρόνος δεν περισσεύει για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα μετά από την Ντόχα όπου πρέπει να επιτευχθούν κάποιοι συμβιβασμοί. Και στο άρθρο 3 το ψήφισμά μας λέει ότι εκφράζουμε κάποια αρκετά σημαντική ανησυχία. Ίσως μπορεί αυτό να ενισχυθεί ως διατύπωση, διότι πραγματικά έχουμε ανησυχίες και τον φόβο ότι ίσως στην Τόχα ε, δεν θα ακουστούν παρά μόνο λόγια και τίποτα επί της ουσίας. Το πρωτόκολλο του Κιώτο πρέπει εκεί επιτέλους να συμφωνηθεί, το είπε η Σάτου Χάση. Χρειαζόμαστε ακαιρεότητα του πρωτοκόλλου και για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα AAUS δεν συνυπολογίζονται. Πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση εσωτερική. Ε, να συζητηθεί το θέμα με την Πολωνία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο Κιώτο 2 και να κουβαλάμε μαζί μας το φορτίο αυτό. Αυτό θα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για τη Ρωσία και την Ουκρανία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί η Κομισιόν ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές ενδιαφέρουσα θα είναι και η διάρκεια, η διάρκεια ισχύως του Κιώτο 2, 5 χρόνια ή 7 χρόνια. Γιατί για την Ένωση το 2020 είναι ευνοϊκό διότι έχουμε στατηγική 2020, έχουμε στόχους 2020, επομένως συμπίπτουν, συμπίπτει το 2020 ως ορίζον και με τους στόχους αυτούς. Βέβαια οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αναμένουν να πούν ότι αν βάλουμε το πλαίσιο στα 7 χρόνια τότε θα πρέπει και οι στόχοι να ανέλθουν. Δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή το τον ίδιο στόχο μείωσης για τα 7 χρόνια όπως για τα 5 χρόνια. Και φοβούμε ότι για το 2020 ο στόχος το 30% έχει χαθεί. Ούτε καν στο δικό μας ψήφισμα δεν αναφέρεται. λέει η επιστήμη ότι θα πρέπει να είναι μεταξύ 25 και 40%. Αυτό το λέμε και το αναμυρικάζουμε. είναι όμως αφηρημένο και δεν είναι δεσμευτικό. Όταν γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε ήδη στο 2012 στο 17,5% μείωση το διοξιδίου του άνθρακος, θα πρέπει να είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να περιλάβει στο κείμενό του ένα υψηλότερο στόχο. Γνωρίζουμε βέβαια πόσο δύσκολο είναι αυτό ε, ακόμη και εδώ στη δική μας Ολομέλεια. Όμως η Επιτροπή Περιβάλλοντος μπορεί να προωθήσει ένα πιο φιλόδοξο στόχο. Συμφωνώ με την Σάντου Χάση ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανεβάσει τον πύχη τότε πολλά κινδυνεύουν να χαθούν. Στην Τόχα θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και το τι σημαίνει χρηματοδότηση. Διότι κάπως είναι ασαφή τα πράγματα, λίγο στα τυφλά προχωρούμε σε ό,τι αφορά καινοτόμε πηγές χρηματοδότησης. Ένας ενδεχόμενος, μια ενδεχόμενη πηγή είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, άλλος είναι ένας ενδεχόμενος φόρος επί της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Πρέπει τα πράγματα όμως να γίνουν πιο συγκεκριμένα. Αλλιώς και μετά το 2012 θα έχουμε το κενό. Εγώ συμφωνώ επίσης με το ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα πρέπει να συμφωνήσει πριν από τη διάσκεψη της Ντόχα και όχι όπως έγινε σε Ντέρμπαν και Κανκούν στη διάρκεια της διάσκεψης και μέσα σε ε, συνεδριάσεις κρίσεως. Ασφαλώς και πρέπει να μιλήσουμε μια φωνή, αλλά αλλιώς δεν ακούγεται η φωνή της Ευρώπης αν δεν είναι ενιαία. Όλες οι χώρες μέλη πρέπει να δείξουν λοιπόν κάποια πειθαρχία, κάποια αυτοπιθαρχία καλύτερα και να επιτευχθεί η συνένεση. Η συνθήκη για το κλίμα που υποτίθεται ότι θα υπογραφεί το 2015 δεν έχει απαραίτητα πολύ χρόνο στη διάθεσή της ακόμα. Δηλαδή δεν είναι και πολύ ο χρόνος από το 12 μέχρι το 2015. και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση ώστε στην Τόχα ήδη να συμφωνηθούν τα βασικότερα, τα πιο θεμελιώδη στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Τελευταία μου παρατήρηση, το Κατάρ προσκάλεσε δεν ξέρω η παρούσα προεδρία τι στάση τηρεί μέχρι τώρα τι κάνει το Κατάρ δηλαδή στα πλαίσια της διεθνούς προστασία του κλίματος. Από την εποχή του Μεξικού ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Προεδρίας. Το ίδιο είδαμε και στην Νότια Αφρική. Με κάποια παράγραφο λοιπόν ίσως πρέπει να ενθαρρύνουμε την επερχόμενη Προεδρία της Διάσκεψης για το Κλίμα να αναλάβει ενεργότερο ρόλο. Ευχαριστώ. Γερμπραντή που αντικαθιστά την κυρία Λεπάζ, η οποία είναι συνεισηγήτρια του εγγράφου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς η συνάδελφος δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα. Η πρώτη μου σκέψη όταν κατάλαβα ότι είχαμε την επόμενη κόπη στο Κατάρ ήταν ότι ίσως είναι ένα παράδειγμα της κοινικής κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις περί κλίματος διεθνώς. Γιατί το Κατάρ είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές κατά στον κόσμο. Και εκεί ακριβώς προσπαθούμε εμείς να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ελπίζω να είναι απλά κινησμός και όχι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί μια προφητεία. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για το τι θα συμβεί στην Τόχα, κυρίως γιατί το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου του Κιώτο θα γίνει μετά την Τόχα. Ωστόσο, έχουμε κάποιους στόχους εκεί. Επειδή κυρίως η του Χάση και ο Τζον Λάινεν ήδη είπαν πολλά σημαντικά πράγματα, δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό όχι μόνο να μιλάμε για ευρωπαϊκή ηγεσία στα διεθνή φόρα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορούμε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από ό,τι ήμασταν τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Ένα από τα στοιχεία που εγώ επαναλαμβάνω εδώ και κάποια χρόνια είναι πότε θα πάψουν οι επιδοτήσεις στην ε, ρήπανση. Το συζητάμε εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουμε φτιάξει κανένα πρόγραμμα δράσης με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα και σταθερά χρονοδιαγράμματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς την Κομισιόν. Πότε ε, θα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό το τομέα. Δεύτερη και τελευταία παρατηρήση είναι ναι, διανύουμε κρίση οικονομική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προωθούμε τις, ε, δεν θα πρέπει να προωθούμε τις επενδύσεις ε, ή τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει στο παρελθόν σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Μέχρι στιγμής έχουμε δεσμεύσει ή πληρώσει μόνο τις 4% ε, των δεσμεύσεων των τελευταίων ετών. <coughs> Ξέρουμε ότι ο λογαριασμός αυξάνεται όταν δεν δρούμε άμεσα. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα μόνο αν δεν ενεργήσουμε άμεσα. Ερώτησή μου προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο φυσικά είναι ως εκ τούτου τι θα κάνουμε ώστε σοβαρά να, να λειτουργήσουν και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλάβουμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πραγματικά έχω αγχωθεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση. Γιατί κάθε φορά που σημειώνεται κάποια πρόοδος στις μετρήσεις και στις παρατηρήσεις, η πρόοδος είναι αρνητική σε σχέση με την ε, σημερινή κατάσταση. Να πω ότι γίνεται μία μελέτη αυτή τη στιγμή για τα, τους παγετώνες της ε, Ανταρκτικής που δείχνει μία ταχύτητα τήξης που είναι δύο με τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτήν που είχε αρχικά υπολογιστεί. Μα τέτοια πράγματα, τέτοιες πτυχές, τέτοια νέα έχουμε τις τελευταίες μέρες και νομίζω λοιπόν πως πρέπει πραγματικά να γίνει, ε, να ξανασκεφτούμε μάλλον εντελώ την κατάσταση. Ακριβώς επειδή λίγα πράγματα όπως η θέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου που δεν έχει σημασία από πού εκπέμπονται γιατί καλύπτουν ολόκληρη την υφήλιο όλα αυτά φωτίζουν αυτή την κατάσταση αλληλεξάρτησης που επικρατεί ανάμεσα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να επικρίνουμε την έννοια της κυριαρχίας εδώ. Γιατί εφόσον είμαστε αλληλεξαρτώμενοι, η ε, κυριαρχία δεν είναι πλέον απόλυτη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αναζητήσουμε βάσεις, ε, βαθύτερες βάσεις για συμφωνίες. Εντάξει η κλιματική διπλωματία, αλλά πιστεύω πως είναι πιο σημαντικό να κατανοήσουμε ποια είναι η βάση που μπορεί να κάνει την κατάσταση να κινηθεί και θα πρέπει να φιλοδοξούμε για περισσότερη κλιματική δικαιοσύνη. Α θυμηθούμε πως εμείς ακόμα δεν δώσαμε πολιτική απάντηση στην ε, δήλωση του Μπαλί για την κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη. Γιατί αυτό είναι το νόημα του όσων πρέπει να κάνουμε. Διότι είμαστε υπεύθυνοι ως έθνη ε, ανεπτυγμένα για ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του αποθέματος ε, των αερίων του θερμοκηπίου που ήδη βρίσκεται στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε αυτό το μέρος της ευθύνης, αυτή την ευθύνη απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κλιματική δικαιοσύνη σημαίνει ακριβώς να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να κατανείμουμε για παράδειγμα τα δικαιώματα εκπομπών με τέτοιο τρόπο ώστε οι ανεπτυγμένες χώρες να είναι αυτές οι οποίες θα φέρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του κόστους. Ακριβώς λόγω της δικής μας ευθύνης για το ήδη υπάρχουν απόθεμα ρήπασης. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να στοχεύσουμε να μην υπάρχουν ε, δωρεάν άδειες εκπομπών παρά μόνο για ένα κομμάτι το οποίο να είναι βιώσιμο. Αν θέλουμε να μειώσουμε στο 1 πέμπτο τουλάχιστον την συγκέντρωση των ε, ε, των αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειώσουμε κατά, ε, με έναν, ένα συντελεστή 5 τις εκπομπές. Το 20% που παραμένει αν είναι βιώσιμο λοιπόν θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των ε, ανθρώπων που ζουν στην υδρόγειο και στις μελλοντικέ γενναίες δωρεάν. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να είναι επιπληρωμή οι άδειες. Με αυτή την έννοια μιλώ για κλιματική δικαιοσύνη, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται αυτό το δικαίωμα των ανθρώπων σε ίση πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και ως εκ τούτου ε, τη δυνατότητα ε, να απορρίπτει κανείς ε, ρήπου στην ατμόσφαιρα είναι ένα από τα δικαιώματα. Βαθιές αλλαγές λοιπόν χρειάζονται εάν θέλουμε πραγματικά οι διαπραγματεύσεις να φτάσουν σε κάποιο αίσιο πέρα. Πιστεύω πως είναι τώρα πια αργά για την Τόχα, αλλά τουλάχιστον μεταξύ μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να λέμε πια παραμύθια και μόνο εάν κάνουμε μια πραγματικά εις βάθος δουλειά υπέρ μιας κλιματικής δικαιοσύνης θα φτάσουμε σε κάποια λύση. Διαφορετικά θα επέλθει η καταστροφή. Ευχαριστώ. Κυρία Κόρολα, ευχαριστώ. Κοιτώντας το ψήφισμα και τα συμπεράσματα, νιώθω ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξο όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ντέρμπαν. Για την μείωση των εκπομπών είναι προφανές ότι η βάση που δημιουργήθηκε στο Ντέρμπαν και το Κιώτο 2 θα είναι κάτι ασήμαντο. Αν δούμε το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα του Τέρμπαν. 27 ευρωπαϊκές χώρες, 10 μικρούς, που εκπέμπουν λίγο δηλαδή. Και άλλες αναπτυγμένες χώρες χωρίς ουσιαστικά υποχρέωση μείωσης. Άρα θα καλύψουμε το 50% των παγκοσμίων εκπομπών. Συνεπώς, το σημείο Β, για παράδειγμα, που λέει ότι το πακέτο Ντέρμπαν έθεσε τα θεμέλια για μελλοντικές δράσεις, εγώ δεν είμαι τόσο φιλόδοξη. Αφού ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, είναι εκτός η Ρωσία, ο Καναδάς και οι, αυτοί που ρηπαίνουν περισσότερο έχουν επιλέξει άλλη προσέγγιση. Το θέμα δεν είναι να βάζουμε οροφές, αλλά να μειώσουμε τις εκπομπές του εξωτερικού του άνθρακα. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν κάνουν τίποτα, είναι ότι έχουν ε, επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την κλιματική πολιτική. Για μένα αυτό ακριβώς είναι μήνυμα αδυναμίας από πλευράς της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι έχουμε ηγετικό ρόλο και ναι, αλλά ε, για το όνομα του Θεού. Leadership σημαίνει ότι εγώ είμαι μπροστά και εσείς ακολουθείτε εμένα. Ας ξεχάσουμε λοιπόν αυτή την ιδέα γιατί δεν ισχύει. Δεν έχουμε δει την Ευρώπη να έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Το σύστημά μας είναι αναποτελεσματικό, είναι ακριβό και δεν ενθαρρύνει τελικά προς την κατεύθυνση που θέλουμε, δηλαδή μείωση των εκπομπών δεν είναι ένα καλό μήνυμα που στέλνουμε στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ξαναδούμε, θα ξανακοιτάξουμε και θα αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας και τη μεθοδολογία μας. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε δύο, λεπτά από εδώ και μπρος, δεν προλαβαίνουμε. Ο Πέτερ Λίζε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συνεισηγητές και συνεισηγήτριες. Σήμερα κειμένο τα αισθήματά μου. Γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της αλλαγής του περιβάλλοντος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πάντως ούτε ορθό, ούτε πολιτικά σκόπιμο να προωθούμε εδώ σενάρια καταστροφής, είτε προς τη μία είτε προ την άλλη κατεύθυνση. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να καταστραφεί, ούτως ή και ούτε επίσης ούτε επίσης σημαίνει ότι άλλα μέρη του κόσμου δεν επιθυμούν να κινητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να προβάλλουμε τέτοια σενάρια ολικής καταστροφής. Δεν είναι υπερβολικά αργά, δεν είναι, ούτε του χρόνου θα είναι υπερβολικά αργά. Απλώς οι λύσεις γίνονται όλο και πιο δαπανηρές, όλο και πιο ακριβές. Και όσο νωρίτερα αρχίσουμε να δουλεύουμε, τόσο λιγότερες θα είναι οι ζημιές που θα υποστούν κυρίως οι φτωχότεροι των φτωχών. Και βεβαίω δεν είμαστε μόνοι μα. Αναφέρομαι κυρίως στην παράγραφο 15, όπου βέβαια αναφερόμαστε στις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές. Θέλω να ρωτήσω όμως και την Κομισιόν, τι ρόλο θα παίξει αυτό στο Ντέρμπαν, όχι στην Τόχα, στην Τόχα διορθώνω. Μπορεί κανείς εκεί να αναμένει υποστήριξη της συμμαχίας της Ντόχα που ήταν οι φτωχότερες χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ο Γιώ Λάινεν αναφέρθηκε πάλι στο 30%. Δεν μας εξυπηρετεί αυτό. Έγιναν τροπολογίες ήδη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη σχετική έκθεση για να κατέλθουμε στο 25% και ίσως χρειαστεί και άλλη μείωση να μην μιλούμε για τα 30%. Να βασιστούμε στον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε τότε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Η κυρία Γιολάντα Χίπνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα η διάγνωση. Η διάγνωση. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για 12-15% των παγκόσμιων ε, αερίων του θερμοκηπίου. Οι μεγάλες ε, χώρες, οι ομάδες χωρών που κάνουν τη μεγάλη ζημιά δεν επιθυμούν να συνεργαστούν. Έχουμε συμφωνήσει να προσπαθήσουμε να μην, ε, υπερβεί η αύξηση θερμοκρασία στους δύο βαθμούς Κελσίου. Η COP17 ήταν επιτυχία. Δεν ήταν αποτυχία, από όσο ξέρω εγώ. Η Πολωνική Προεδρία λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορηθεί για την έλλειψη μεγαλύτερης επιτυχίας. Μπορείτε να υπογράψετε ό,τι θέλετε στις, δια, αλλά αν δεν υποστηρίξουν οι μεγάλες χώρες παραγωγής διοξιδίων του άνθρακα, όπως η Ινδία, η Κίνα, οι Ενωμένε Πολιτείε, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσετε. Το 20% είναι ρεαλιστική προσέγγιση. Οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ότι μπορούμε να επιτύχουμε και το 25%. Υπάρχει κίνδυνος ότι οι εκπομπές θα εξαχθούν σε άλλες χώρες, χώρες οι οποίες δεν επιθυμούν να συνυπογράψουν τις ε, αποφάσεις μας. Τότε θα σηκωθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα πάει αλλού. Και αυτό που θα έχουμε εμείς θα είναι η υψηλότερη ανεργία. Υπενθυμίζω στον συνάδελφό μου από τη Δανία που κατηγόρησε τόσο την Πολωνική Προεδρία ότι η Δανία δεν μας εκπροσώπησε καλά την περιοχή Σέγγεν δηλαδή, όπως το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Σούλτς. Σήμερα το θέμα είναι η προπαρασκευή της διάσκεψης COP18 και όχι αξιολόγηση των πεπραγμένων διαφόρων προεδριών. Το υπενθυμίζω αυτό σε όλους και όλους τους συναδέλφους. Η Μαρίτα Ούλσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως η Προεδρία παίζει ένα ρόλο. Και η Πολωνία θα μπορούσε να είχε επιτύχει περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Άρχισε βέβαια η υπόθεση ε, με την προπαρασκευή στην Κοπενχάγη και αυτό έγινε υπό Σουηδική Προεδρία. Και μετά είχε ακολουθήσει η Δανέζικη. Και η Δανέζικη και η Σουηδική Προεδρία κάνανε μεγάλα λάθη στη διάρκεια της συνδιάσκεψης. Όλα αυτά βέβαια έχουν σχέση και με το τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε και με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί, που οδήγησε τελικά ο πρόεδρος Ομπάμα να μην μπορέσει να επιτύχει τα όσα αναμένονταν από αυτόν. Και εμείς όμως κάναμε ως προεδρίες λάθη και αντιμετωπίσαμε μετά πολύ γρήγορα σοβαρές συγκρούσεις με άλλα τμήματα του κόσμου. Με λίγα λόγια όλοι κάνουμε λάθη. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να φροντίσουμε στο μέλλον να κάνουμε λιγότερα σφάλματα και να προχωρήσουμε, διότι έχουμε ένα φιλόδοξο επίπεδο το οποίο αναγκαστήκαμε να μειώσουμε σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, αύξηση της ε, θερμοκρασίας. πρέπει να ακολουθήσουμε ρεαλιστικούς στόχους. Η Σάτου Χάση και οι άλλοι συνάδελφοι που μίλησαν όπως η Ολάινεν έχουν δίκιο. Η συνέχιση του Κιώτο πρέπει για μας να είναι κύριο, κύριο στόχος και το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να εκφράζουμε μόνο ευχές πρέπει να συμφωνήσουμε και για το ποια πράγματα θα αναλάβουμε. Δηλαδή, πρέπει να είναι πρώτη της προτεραιότητας η χρηματοδότηση και το κοιότο και χρειαζόμαστε στέρεα προετοιμασία σε συνεργασία με την Κομισιόν πριν από τη διάσκεψη, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι στη διάσκεψη. Χρειαζόμαστε έναν κατάλογο με πράγματα που πρέπει να γίνουν Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είμαι από τους υπογράφοντες, λέει ο κύριος Ούσκι, αλλά δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο. Και δεν είμαι και ικανοποιημένος από την πρόοδο. Στον Παλί. Όλοι επέστρεφαν από το Παλί λέγοντας ότι ναι, όλα είναι ξεκάθαρα και ότι αρκούσε πια να γίνει μια ακόμα μόνο διάσκεψη ώστε να φτάσουμε σε μια σφαιρική συμφωνία. Η διάσκεψη επόμενη αυτή της, της Κανκούν κυρίως ήταν ε, σχεδόν τελείω αποτυχημένη. Η μόνη επιτυχία ήταν ότι έγινε δεκτή μια δήλωση για τη συνέχιση των, ε, των διαπραγματεύσεων. Και τώρα Εμεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και δεν μιλάω μόνο για το Κοινοβούλιο, μιλάω για το σύνολο της Ένωση. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε, έχουμε υιοθετήσει ένα, μέτρο, ένα πακέτο μέτρων, έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών, έχουμε, στηρίζουμε τις σύγχρονες τεχνολογίε αποθήκευση άνθρακα και έπειτα αν δούμε υπάρχουν άλλοι που εκπέμπουν αέριο του θερμοκηπίου σε, με, σε τεράστιους όγκους όπως η Κίνα και αυξάνει συνέχεια μάλιστα τις εκπομπές της. Το αδύναμο σημείο λοιπόν της σημερινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς ε, ε, η διπλωματία η περιβαλλοντική διπλωματία. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε αρκετά εργαλεία, δεν έχουμε αρκετά ιδέες δυνατότητες να, πα, να, να διεκδικήσουμε και να προωθήσουμε τα σχέδιά μας. θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή Διεθνούς Στρατηγικής Κλίματος στη Γενική Διεύθυνση, στη Διεύθυνση Κλίματος μάλλον. Έχουν κάνει ερωτήσεις οι συναδελφοί μου και παρακαλώ να τις σχολιάσετε και κυρίως ό,τι αφορά την εφαρμογή. Καμιά φορά εδώ στην Ευρώπη έχουμε την ιδιότητα να επενούμε πάρα πολύ μια διάσκεψη ή να την καταδικάζουμε ως απόλυτη αποτυχία. Σαν να μην υπάρχει τίποτα ενδιάμεσα. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Και μετά από την διάσκεψη, τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς σκέπτεται ότι ε, ε, ε, πώς έγινε δηλαδή η, η εργασία εκεί στη διάσκεψη και αυτό βέβαια να το λάβουμε υπόψη και στις εργασίες μας και μια παράκληση αν και είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Και η παράκλησή μας είναι να είναι πλήρης η συμμετοχή της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα θεσμικά. Εφόσον ένα κοινοβούλιο καταβάλει προσπάθεια και εγκύπτει στην μελέτη του θέματος, γνωρίζω βεβαίως ότι έχουμε καθεστώς παρατηρητού, δεν είμαστε μέλη. Έχουμε, όπως είπα, καθιστός παρατηρητού και αυτό πρέπει να το προσέξουν οι συναδελφοί μου. Για την εφαρμογή μετά όμως, χρειάζεστε τους 70 συναδέλφους της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος, καθώς τους 70 συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και τους 700 ε, ευρωβουλευτές. Και για να περάσει και στην κοινωνία. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε μια αξιοπρεπή συμμετοχή μας στην ε, διάσκεψη για το κλίμα. Αυτό θα είναι και από, ένα από τα χέγγια της επιτυχίας, αν θέλετε, για το τι φορά. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια για την προετοιμασία της Δόχα. Όπως όλοι αναγνωρίζουν, η ΔΟΧΑ δεν θα αποτελέσει ένα, μια πολύ σημαντική αλλαγή στα όσα κάνουμε μέχρι τώρα αλλά πρέπει να προχωρήσουν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Πέντε πράγματα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το πρωτόκολλο του Κιώτου και τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης που πρέπει να ξεκινήσει 1η Ιανουαρίου του 2013. Πρέπει επίσης να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για το πρόγραμμα δράσης πάλι, κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει νέους μηχανισμούς στην αγορά, αλλά και το θέμα της εφαρμογής του μπαλί. Ε, πρέπει επίσης να δούμε τι έχουν υποσχεθεί η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι εταίροι μας δηλαδή, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τη συμφωνία και να δούμε και να φροντίσουμε να τρίσουν τις δεσμεύσεις τους. Το δεύτερο είναι η πλατφόρμα Durban. Εδώ το πιο σημαντικό είναι να πλαισιώσουμε τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις για την επόμενη τριετία και να πετύχουμε συνένεση από αυτού. Είναι αλήθεια ότι στη Βόνη δεν ε, πετύχαμε πολλά. Αγωνιστήκαμε για την σε διάταξη, αλλά οι συζητήσεις στην Μπαγκόγκ ήταν επικοδομητικές από αυτού. Και ήδη βλέπουμε τη μορφή του προγράμματος δράσης, ιδιαίτερα για το έτος 2013. Το τέταρτο είναι ε, το χάσμα φιλοδοξιών. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Είναι αλήθεια. Μετά το Ντέρμπαν δεν ε, είχαμε μπει στο δρόμο να πετύχουμε τους δύο βαθμούς, άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα εδώ. Επειδή όλοι αναγνωρίζουν τις πολιτικές και γεωπολιτικές πραγματικότητες, θέλοντας να μειώσουμε το χάσμα, ιδιαίτερα από πλευρά των ΗΠΑ τι ισχύει. Δεν υπάρχει μια ε, κυβέρνηση η οποία θα θέλει να πετύχει το στόχο, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τηρήσει τις δεσμεύσεις της η Αμερική. Όμως συζητούμε από τις πλευρές εκείνες που ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα, που είναι πάνω από 200 χώρες, ούτε στο Κανκούν, ούτε αλλού, να έρθουν και να προχωρήσουν προς τους στόχους. Το Κατάρ πράγματι είναι μία από αυτές τις χώρες που δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση σε διεθνέ επίπεδο για κλιματικές αλλαγέ. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν το έχουν κάνει. Η Μαλαισία, η Ταϊλανδία, το Βιετνάμ, Αναδυόμενε οικονομίες Επίση μπορεί να κάνουν κάτι για το κλίμα, αλλά σε διεθνέ επίπεδο δεν έχουν δεσμευτεί. Το άλλο που πρέπει να δούμε είναι συμπληρωματικά μέτρα. Ένα πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το phasing out, δηλαδή την σταδιακή μείωση των ε, ενισχύσεων. Αν αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να τη διαβρύνουμε και να συμπεριληφθούν στην πρωτοβουλία αυτή και άλλες χώρες, αυτό θα βοηθούσε πράγματι να μειώσουμε παρατέρω τις εκπομπές. Ή έπειτα υπάρχουν και άλλες για το μαύρο άνθρακα εκπομπές. Τι κάνουμε με αυτό ή για άλλα αέρια ή να δούμε πώς μπορούμε να επιτεχύνουμε τη δράση μας κατά της ε, αποψήλωσης των δασών. Δεν λέω ότι είμαι αισιόδοξο πως θα ολοκληρωθούν όλα αυτά, αλλά μη τι άλλο πιστεύω ότι μπορούμε κάτι να προχωρήσουμε. Το πέμπτο είναι το θέμα των, ε, της οικονομίας ε, του κλίματος. Για το 2012 πρέπει να είναι ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν τα χρήματα για το 2012 ώστε 100% να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στην Κοπεχάγη. Αλλά πρέπει να δώσουμε και κάποια προοπτική για το τι θα γίνει στη συνέχεια, το 2013 και το 2014 δηλαδή. Άρα και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει, γιατί εσείς θα αποφασίσετε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013 σε λίγες εβδομάδες. Αν λοιπόν στείλετε ένα μήνυμα και για ε, τα χρήματα που θα πάνε στο κλίμα, αυτό θα βοηθούσε την Τόχα. Τώρα αναφερθήκατε και σε δύο ειδικά ζητήματα. Το πρώτο είναι τα αποθέματα κατά κάποιο τρόπο ρήπανσης μετά το Κιώτο. Όντως αυτό είναι ένα θέμα που διχάζει τις χώρες μέλη. Και όσον αφορά την ε, περιβαλλοντική κυριότητα όντως είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί στην Τόχα. Όμως θέλω να σας υπενθυμίσω εδώ κάτι και αυτό είναι ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουμε απόφαση το 2008 όταν ε, εγκρίθηκε το πακέτο ενέργειας και κλίματος που έλεγε ότι αυτά τα επιπλέον AAUs ε, είναι για να τηρήσουν τα κράτη τις δικές τους δεσμεύσεις υπό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άρα λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τιμήσαμε τις ε, υποχρεώσεις μας όσον αφορά δηλαδή το δικό μας πακέτο του 20%. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον ε, μηχανισμό ε, καθαρών, ε, καθαρής ανάπτυξης. Εδώ ο μηχανισμός δεν είναι ακριβώς η συνέχιση των CDM την επόμενη περίοδο. Έχουμε Όντω μια κακή ισορροπία για τα μα όσον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά. Η αγορά δυστυχώ έχει γεμίσει με πιστώσει όσον αφορά τα δικαιώματα ρήπανση. Χωρί να υπάρχει όμω ε, ζήτηση παρετέρα, Άρα, λοιπόν οι τιμέ ε, μειώνονται. Άρα το θέμα είναι να κοιτάξουμε την ισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά. Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ξέρετε ότι εμείς το κοιτάμε αυτό στα πλαίσια της εμπορίας δικαιωμάτων ρήπανσης, αλλά και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί να πάρει κάποια απόφαση τους επόμενους μήνες για να αποκατασταθεί η ισορροπία αυτή ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Μια άλλη ερώτηση που κάνατε είναι για την περιβαλλοντική διπλωματία. όντω είναι κάτι πολύ σημαντικό και το δεύτερο εξάμεινο κάθε χρονιάς παίρνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Μάλιστα, μέσα στη χρονιά αυτή, προετοιμάζοντα τη διάσκεψη τη Ντόχα, έχει γίνει ελάχιστη πρόοδο. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση στη ε, Νέα Υόρκη από τις μεγάλες οικονομίες και εμείς από Ευρωπαϊκή Ένωση θα συναντηθούμε με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε μια παρασκευαστική συνάντηση στη Σεούλ στην ε, Κορέα. Άρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι ακόμα παραπάνω και αν ε, η Προεδρία του Κατάρ θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να το θίξουμε. Αλλά τουλάχιστον Κάτι θα συζητήσουμε με τους φίλους από το Κατάρ. Και επίσης η ΑΕΣ δραστηριοποιείται όσον αφορά την παραλωτική διπλωματία. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα κυρίως μετά το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, όπου το Συμβούλιο εκεί θα αποφασίσει τη διαπραγματευτική εντολή και θα είναι ξεκάθαρο πια για τους εταίρους μας το τι θέλουμε να πετύχουμε εμείς στην Τόχα και ποια κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Τέλος. Έρχομαι και στο θέμα που πάντα συζητάμε κάθε φορά που μιλάμε για την προετοιμασία της διάσκεψης, δηλαδή ποια θα είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη δικιά μου την πλευρά, από πλευρά τη Επιτροπής δηλαδή, Πρέπει να σας πω ότι εμεί θα συνεχίσουμε να θέλουμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Εσείς θα ενημερώνεστε καθημερινά από εμά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, και από τους Επιτρόπους. Υπάρχει η υπόσχεση. Γνωρίζουμε ότι τίθεται κάποια θεσμικά ζητήματα όσον αφορά το Συμβούλιο. Μπορώ όμω να σα διαβεβαιώσω από την πλευρά τη επιτροπή τουλάχιστον ότι εμεί θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να σας ενημερώνουμε για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε τον ε, ρόλο σας μετά όσον αφορά την εφαρμογή των ε, διαπραγματεύσεων όταν αρχίσει η δεύτερη περίοδος για την επικύρωση. Συνεπώς η πρόταση αυτή θα γίνει και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο. Άρα θα έχετε να παίξετε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Στις 26 Ενάτου, 12 το μεσημέρι, λήγει η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. θα ψηφίσουμε στις 6 Δεκάτου εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον Νοέμβριο του 2012 θα καταλήξει η έκθεση σε ψηφοφορία στην περίοδο συνόδου. Έχουμε τώρα προφορικές ερωτήσεις για Συμβούλιο και Κομισιόν. Όποιοι συμφωνούν παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι. Παρακαλούνται να γύρουν την χείρα. Ομόφωνα λοιπόν, καλά. Προχωρούμε λοιπόν. με ρώτησαν, με, με επέβαλε TV 24. Είναι τα κανάλια που βρίσκονται εδώ. Τον ήχο μπορούν να λάβουν οι κάμερες από το web stream, από το διαδίκτυο, διότι μεταδίδεται η συνεδρίαση από το διαδίκτυο. Εδώ έληξε το θέμα 4 και ακολουθεί το 5, Καρδίνη. Και το λόγο λαμβάνει η κυρία Ελιζαμπέτα Γκαρδίνη, η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομη γιατί δεν έμεινε και πολλής χρόνος για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα τη σημερινή διάταξης. Άρα λοιπόν δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Ήθελα μόνο να θυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε εδώ μια προσπάθεια πολύ κοντά στις ευαισθησίες των Ευρωπαίων πολιτών και κατά τη γνώμη μου το έγγραφο το οποίο επέβαλε η Κομισιόν είναι εξαιρετικό σημείο εκκίνησης γιατί η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών ε, που δεν, ανησυχίες που δεν έχουν ξεπεραστεί τελείως στο Συμβούλιο από όσο έχω καταλάβει από διάφορα μηνύματα. Σήμερα, ε, βέβαια πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίου μήνε με τη Δανεική Προεδρία και με την Κυπριακή Προεδρία έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με την Επιτροπή κάνουμε εξαιρετική νομίζω δουλειά. Τώρα χρειαζόμαστε ένα κοινοβούλιο το οποίο κατά παράδεση θα δείξει την βούληση και το θάρρος για να κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά και να εμβαθύνει με μια συζήτηση, μια διευκρίνηση τα σημεία τα οποία μπορεί να ανησυχούν ακόμα κάποια κράτη-μέλη. Τη δική μου δουλειά δεν χρειάζεται τώρα να σας την αναλύσω γιατί ήδη στο σχέδιο έκθεσης είναι σαφής η θέση μου και η σκέψη μου. Εμεί χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο μέσο το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, φυσικές καταστροφές και ακούσαμε και για τις κλιματικές αλλαγές, για τη συχνότητα και την ένταση αυτών των φυσικών καταστροφών που δυστυχώς θα είναι διαρκώς ανησυχητική, είτε πρόκειται για καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο. Παναλαμβάνω λοιπόν, οι στατιστικές δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν περισσότερη Ευρώπη στη διαχείριση των καταστροφών αυτών και να καθησυχάζουμε τα κράτη ότι αυτή η αλληλεγγύη συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την επικουρικότητα, ότι η πολιτική προστασία είναι απόλυτη αρμοδιότητα και εθνικού επίπεδου και περιφερειακού επίπεδου εκεί όπου υπάρχει η περιφερειακή αρμοδιότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό και δυνατότητες καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας μέσω του συνδυασμού αυτών. Έχουμε Μάλλον χρειαζόμαστε την αύξηση και την πρόοδο σε, αυτές, σε αυτό την υπόθεση. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει πολλά σε επίπεδο κομισιών και κρατομελών. Η πολιτική προστασία και ο συντονισμό, η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη και τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, έχει βελτιωθεί. Είδαμε και την εμπειρία φέτος το καλοκαίρι για ορισμένα πιλωτικά πρόγραμμα που έχουν βασιστεί στους ε, κανόνες, αυτό που θα αποτελέσουν τους κανόνες ε, αυτής ε, της εφαρμογής της πολιτικής προστασίας και που λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο τώρα εδώ στο Κοινοβούλιο είναι να παίξουμε ένα συγκεκριμένο και αποφασιστικό ρόλο ώστε όλοι μαζί να δώσουμε την απάντηση που αναμένουν οι πολίτες. Αυτά έχω να πω για να μπορέσουν να πάρουν το λόγο και οι συνάδελφοι και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε και με προσωπικές επαφές για όποιον το επιθυμεί. um Θέλω να αρχίσω στις 10.30 τις ψηφοφορίες που θα είναι μαραθώνιος ψηφοφοριών σήμερα, γι' αυτό θα παρακαλέσω πρώτα η σκιώδηση συγγήτρια, η κυρία Εστέλα, η Ρεμπέκα Τέλερ, Kollege Ματίας, Anna Ροσπαχ Oreste Rossi και τόν dann die Kollegin Sommer. Αυτά είναι τα ονόματα των εγγεγραμμένων. Ως σκιώδεις ηγητές έχουν πρώτοι το λόγο και μετά οι υπόλοιποι. Μετά Μπούβιν και Ζέιμπαχ. Σνέλχαρτ επίσης. Ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα ο χρόνος αγορεύσεως. Εκτός εάν δεχθεί ο εισηγητής να ξανασυζητήσουμε αν θεωρήσει δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω συζητήσεων. Αλλιώς θα πω 1,5 λεπτό και αρχίζουμε αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ήδη είπαμε και το επαναλαμβάνω ότι είναι πρόσδεκτη αυτή η πρόταση της Κομισιόν γιατί η συχνότητα των καταστροφών παγκοσμίως ε, αυξάνεται με τεράστιες ζημιές ε, όσον αφορά τόσο τα θύματα όσο και τις οικονομικές ε, ζημιές για πόλεις. Γι' αυτό και θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε πολιτικές πρόληψεις και να προβλέψουμε και έναν μηχανισμό διαχείρισης των καταστροφών και μια ολοκληρωμένη δυνατότητα ανταπόκριση από πλευρά των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση τη Κομισιόν προχωρεί στην κατεύθυνση τη απλοποίηση, τη ευελιξία και τη αποτελεσματικότητα, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Ήθελα να σας αναφέρω το παράδειγμα του προγράμματος πιλότου για την αποκατάσταση μάλλον συγγνώμη, για την δημιουργία ενός ε, σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ε, επιδεινώνεται από τις ε, αντίξωες κλιματικές συνθήκες που και κάποιες φορές πλήττουν ταυτόχρονα διάφορα κράτη-μέλη, έτσι τις δυσκολίες και τις δυνατότητες αλληλοβοήθειας, πράγμα το οποίο ε, δικαιολογεί την ύπαρξη ενός επιπλέον σώματος που θα στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δημιουργήθηκε έτσι ώστε μια καταστροφή μεγάλων διαστάσεων να μπορεί να αντιμετωπιστεί από το κράτος μέλος που την αντιμετωπίζει και, ε, και να μπορεί αυτό το κράτος να βοηθηθεί όταν δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του μόνο του. Για να κλείσω να πω ότι λυπούμεθα που στο Συμβούλιο υπάρχει μη ανασχετική πλειοψηφία, ε, μειοψηφία με συγχωρείτε, και ότι στηρίζονται στο δίθεν ε, κριτήριο της επικουρικότητας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι υπέρ μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ε, για την ε, προστασία μειώνονται έτσι κίνδυνοι και η συνεργασία ανάμεσα των κρατών μελών για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ευχαριστώ πολύ. Τέιλορ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Έκθεση μάλλον. Ναι. Έρχομαι κι εγώ από μια εκλογική περιφέρεια που έχει πληγεί από τέτοιες καταστροφές. Η απροθυμία του Συμβουλίου βέβαια μας προβληματίζει. Πιστεύω όμως ότι οι τροπολογίες, η ένα για παράδειγμα θα βοηθήσει περισσότερο, οι δύο που αναφέρεται στη εθελοντική εργασία θα ήθελα να στηρίξω και μια άλλη εξέλιξη. Αυτή είναι η πρόταση στο άρθρο 5 της κυρίας Γκαρδίνη για την συγκρισιμότητα όταν μιλάμε για τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει στην νομοθεσία, οπότε θα ήθελα να δημιουργηθούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές γι' αυτό. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι τομείς όπου θα ήθελα βελτίωση το θέμα της εθελοντικής ε, βοήθειας που θα πρέπει όντως να παραμείνει σε εθελοντική βάση, αλλά τα κράτη-μέλη θα έπρεπε αν μη τι άλλο να μας εξηγήσουν αν ε, δεν το θέλουν, γιατί μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω τέτοιους λόγους να μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Η ανταπόκριση πρέπει να είναι επίσης πιο ισχυρή και τέλος θα ήθελα να δω τις οικονομικές προδιαγραφές και το θέμα της ενίσχυσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Χάση. Α, όχι, δεν είναι εδώ. Ο Ματίας, Άννα Ρόσπαχ. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Δέχομαι την βασική αρχή που λέει ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε τη διαχείριση κινδύνου στην αναλυτική μας βάση. Υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις για την επικουρικότητα όσον αφορά αυτή την πρόταση. Όμως εμείς δεχόμαστε τις τροπολογίες της συγκήτριας που υπογραμμίζουν την καταρχήν ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να την εκχωρεί στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δηλαδή πρέπει να την έχουν τελικά και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το άρθρο 196 τη Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει την προστασία ε, του πολίτη για να σαν επικουρική στήριξη προς τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση από τα κράτη-μέλη και Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τόσο αναφέρονται στο άρθρο 196. Επίσης τα κράτη-μέλη πρέπει τον σχεδιασμό τους να τον ε, δίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχει και υποχρέωση εντοπισμού εκ των προτέρων εμπειρογνωμόνων, ειδικών δηλαδή, που θα ασχολούνται με το θέμα αυτό. Το άρθρο 9 αναφέρεται και σε δυνατότητα έκτακτης αντίδρασης από πλευράς ε, των χωρών μελών. Ναι, Μπορεί να πρέπει να υπάρχει συλλογικά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά από την άλλη μεριά αυτή πρέπει να ορίζεται πολύ συγκεκριμένα. Και δεν θα πρέπει να έχει το θέμα αυτό δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ούτε μπορούμε να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη μεταξύ τους αν θέλουν να συνεργάζονται. Η ειδική μας ομάδα πιστεύει ότι η αρμοδιότητα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν για μας ανάμειξη της Ευρώπης σε εθνικό επίπεδο. Ενώ από την άλλη μεριά και το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσε να δράσει. Γι' αυτό λοιπόν και θα καταθέσουμε και το Ευχαριστώ κύριε Ρόσπαχ. Υπενθυμίζω σε όλους και όλους ότι στις 10 και 30 αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Και τι χρειάζεται για την ψηφοφορία, την κάρτα σας. όποιο την ξέχασε ίσως σήμερα το πρωί, ας φροντίσει τώρα στα επόμενα 5-10 λεπτά να την ανακτήσει. Η κυρία Ζόμερ, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Και μετά ο κύριος Γιούβιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι την βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση θεομηνιών και άλλων φυσικών καταστροφών φέρουν οι χώρες μέλη. Ο ρόλος της Ευρώπης είναι συντονιστικός και υποστήριξης. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίζει αυτό περισσότερο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, για παράδειγμα, ότι η ευθύνη των χωρών μελών είναι να διαθέτουν επαρκή ικανότητα. Τα κενά δεν μπορούν να τα κλείνουν οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες οι χώρες μέλη είναι υπεύθυνε. Δύο θέματα που δεν λαμβάνει υπόψη στο κείμενό της κ. Γκαρντίνη, άρθρο 6, η εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης των κινδύνων, ναι μεν, αλλά όχι εναρμόνιση. Να μην υπάρξει εναρμόνιση. Ούτε τα σχέδια αυτά να χρησιμοποιηθούν ως βάση για διευρωπαϊκή capacity building. Για το άρθρο 11 μιλεί για ένα θελοντικό pool των ικανοτήτων και οι πόροι, εφόσον έχουν δηλωθεί από τις χώρες μέλη, να προκύπτει από την δήλωση αυτή υποχρέωση για να διαθέτουν τους πόρους αυτούς. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να το αποδεχτώ. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες οι ίδιες που θα αποφασίσουν εάν θα διαθέσουν πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή όχι. Η οικειοθελής δήλωση ύπαρξης ε, των μέσων αυτών, ναι, αλλά όχι υποχρέωση χορήγησής τους. Οι χώρες μέλη, όπως είπα, οι ίδιες είναι αυτές που θα αποφασίσουν τι είδους βοήθεια θα διαθέσουν, χωρίς κανένα εξαναγκασμό είτε από την Κομισιόν ή από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και την Κομισιόν ε, για τις προτάσεις αυτές. Δεν θα πρέπει να αναδιπλωθούμε σε εθνικές ε, αντιδράσεις, θα πρέπει να πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού επέδου. Για τεχνικά παρατηρήσεις έχω να κάνω, κυρία Εισηγήτρια. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτήν την έκθεση λέγοντας ότι οι δυνατότητες οι ευρωπαϊκές θα μπορούσαν να βασίζονται και στις υπερπεριφερειακές ε, τις περιοχές της Ένωσης και στα υπερπότια ε, εδάφη της Ένωσης. Είναι ένα του. Και έπειτα να καταλάβει και ο ευρωπαϊκός κόσμος ότι ε, δεσμεύεται σε μια συλλογική προσπάθεια και αυτή την έννοια έχει αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική ε, ε, το σώμα να κάνουν σπουδαία πράγματα μαζί έτσι οι άνθρωποι ε, μαθαίνουν να ανήκουν σε μια ομάδα δηλαδή στον ευρωπαϊκό λαό κατά τα άλλα πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι ένα βήμα θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε προς, και όχι να το ελαχιστοποιήσουμε ένα βήμα προς το ευρωπαϊκό έθνος Ευχαριστώ την εισηγήτρια που νομίζω ότι έχει συντάξει κείμενο ισορροπημένο. Βεβαίως την αρμοδιότητα διατηρούν οι χώρες μέλη. Νομίζω όμως ότι όλοι φέρουμε την ευθύνη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει κάποια διαλειτουργικότητα των συστημάτων διάσωσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από εμάς τι είδους Ευρώπη είναι αυτή αν δεν τα καταφέρουμε σε μια χώρα μέλος όπου σημειώνεται μια μεγάλη κρίση να μην είναι δυνατόν να αλληλοϊποστηριχτούμε. Είναι λοιπόν σωστό και ορθό στο ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε την απαραίτητη ε, προσπάθεια συντονισμού και βεβαίω να με μένα από τους δε με βέλτιστες πρακτικές. Στο Ευρωβαρόμετρο βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών θεωρείται μαζί με τη σταθερότητα του ευρώ από τα πρώτη στα θέματα προτεραιότητας από τους ε, πολίτες. Ζητώ λοιπόν και εγώ από τις χώρες μέλη να φτιάξουν ακόμα ε, περισσότερο συντονισμό και νομίζω ότι η Ελιζαπέτα Καρδίνη σωστά τα λέει. Σνέλ Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω και εγώ την εισηγήτρια, όπως και οι άλλοι. Σωστό, είναι και καλή η έκθεσή της, αλλά υπενθυμίζω ότι ε, εδώ και 10-15 χρόνια μιλούμε για κοινέ επιχειρήσεις αντιμετώπισης θεομηνιών στην Ευρώπη. Έχουμε διατυπώσει στόχους, έχουμε συντάξει έγγραφα, άρα σπανιότατα γίνονται κοινέ επιχειρήσεις. Εν μέρη βέβαια σε διμερές επίπεδο μετά από συνεννοήσεις μεταξύ χωρών μελών η Κομισιόν προσπαθεί ξανά και ξανά να δώσει ένα πλαίσιο. Εγώ το θεωρώ σωστό. Ουδής αμφισβητεί ότι η προστασία, η πολιτική προστασία πρέπει να είναι στα χέρια των χωρών μελών. Αλλά όταν, αν φτιάξουμε, όταν φτιάξουμε ένα επιτελείο στην Κομισιόν που να προχωρήσει στο συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης των καταστροφών θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να ζητηθεί από τις χώρες μέλη να διαθέσουν πόρους τους οποίους, ε, οποίους έχουν. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα, της χρηματοδότησης. Το κείμενο εδώ μου φαίνεται πολύ χαλαρό. Λέει ότι η συγχρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%, καμιά φορά και στο 100%. Εάν δρούν πλείονες χώρες, τότε η μία είναι, μία είναι αυτή που χρειάζεται να το ζητήσει. Πρέπει να είναι σαφής ή διατυπώσει εδώ. Δηλαδή ποιε δράσεις χρηματοδοτούνται στο 100% πρέπει να είναι αυτές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αλλιώ η γραφειοκρατία θα είναι σημαντική. Ευχαριστώ, Σνέρχαρτ η εισηγήτρια πολύ σύντομα και μετά προχωρούμε αμέσω στην ψηφοφορία. Όλοι παρακαλώ να ελέγξετε αν έχετε τις κάρτες σας. Κυρία Γκαρντίνη, σύντομα. Σα ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να εμβαθύνουμε εδώ στην Επιτροπή περισσότερο για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Και θα συνεχίσουμε τύπως την ε, δουλειά μας όπως το κάναμε και τους τελευταίους μήνες, κυρίως για να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να το μεταθέσουμε αν είχαμε καθυστερήσει και εδώ. Ε, εγώ πιστεύω πως όλες οι προτάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι είναι προτάσεις ε, ε, με στόχο να εμβαθύνουμε, να υποκατασταθμίσουμε και να συνεχίσουμε να προχωρούμε προς την ίδια κατεύθυνση που προτείνει η Κομισιόν. Το μόνο που θα Μα ανησυχούσε ήταν να μένουμε στο status quo. Αν έλεγε κάποιος, δεν το είπε κανείς, γιατί ακριβώς το status quo δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Σας ευχαριστώ όλους και νομίζω πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με πολύ καρποφόρο τρόπο τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 2 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. 5 και 6 Νοεμβρίου θα γίνει συζήτηση εδώ στην Επιτροπή ΕΝΒΗ και 28-29 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Στην Ολομέλεια θα καταλήξει κατά πάσα πιθανότητα η έκθεση το, τον Ιανουάριο του 2013. Προχωρούμε ευθύ αμέσω τώρα στις ε, ψηφοφορίες. Έχουμε το θέμα 6 λοιπόν, έκθεση Παλέκης, μετά Σόνικ, μετά Κάλινμπαχ, Γιόργενσεν, Ματίας και Χάουκ, η απαλλαγή. Αυτά θα ψηφίσουμε. Επομένως τώρα γνωρίζετε και την σειρά. Αρχίζουμε. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Παλέτσκης που είναι παρόν. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 64. Υπέρ, κατά. Αποχές. Θα προχωρήσουμε σε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 64. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Υπέρ 24, κατά 23. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά. Το αποτέλεσμα προηγουμένως ήταν 24 υπέρ 23 κατά, λέει ο Τώρα, τροπολογία 14 κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτουν ορισμένες. Συνεχίζουμε με την 16 υπέρ. Κατά Ας το επαναλάβουμε. Υπέρ. Υπέρ της 16. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο που είναι ταυτόσιμες τώρα. 89 και 69 ή μάλλον 96 ε, δεκτές 19 τώρα συγγνώμη 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 εκπίπτει Καλά. Επαλήθευση της 21 ηλεκτρονική. Ψηφίσατε. Πέρας. Υπέρ 32, 25 κατά. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονικά λοιπόν. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. 30 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαλήθευση. ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Η σοσιαλδημοκρατική ομάδα έχει δύο παραπάνω. Ψηφίζουν δύο παραπάνω. Παρακαλώ δύο να αφαιρέσουν τις κάρτες. Ένας ακόμη λέτε. Ξανακάνουμε την ε, ψηφοφορία για την 23. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. 30 υπέρ, 25 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 31 υπέρ 27 κατά. 94 υπέρ. κατά, αποχές, ίδια πλειοψηφία. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, κατά, αποχές, απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 ε, κατά τμήματα σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επίσης 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 του του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη τροπολογία 3 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 4. Κόντς 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Consolidated 5. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκπίπτει η 31 που έχει περιληφθεί, έχει καλυφθεί μάλλον με την ε, ενοποιημένη. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 32 του συγγήτου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30, όχι λέει ο πρόεδρος, 120. Α, την ψηφίσαμε. Καλά. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται αυτή ενοποιημένη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 ως προσθήκη είδατε 124 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 36 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. για την 36 λέει υπέρ, κατά. Τριάντα υπέρ, κατά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 Κατά. Αποχές. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ο συσχετισμός των δυνάμεων. Ας τον ελέγξουμε ωστόσο ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, το Λαϊκό Κόμμα έχει έναν παραπάνω. Μία ψήφο παραπάνω θα, από τις δικαιοτητες θα πρέπει να αποσυρθεί μια κάρτα. 29 υπέρ, 33 κατά. Απορρίφθηκε επομένω. Ενοποιημένη τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. Ενοποιημένη 7. 7. Ενοποιημένη 7 γίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. 33 υπέρ 28 κατά. Να με πιστεύετε όταν σας λέω το αποτέλεσμα. 137 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση δεν είναι τόσο ξεκάθαρο από το Προεδρείο. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. 27 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 και 147 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές συγγνώμη 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 και 203 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 48. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 59 υπέρ. Καμία κατά και καμία αποχή. Το ίδιο να δείχνετε και τις επόμενες φορές, δηλαδή καθαρά. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 188 υπέρ, Κατά. Χρειάζεται επαλήθευση. Δεν είναι τόσο σαφέ το αποτέλεσμα. 188 λοιπόν. Επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Το Λαϊκό Κόμμα. Μία κάρτα παραπάνω. Καλά λοιπόν. Πέρασε. 38 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193 έχει ζητηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 32 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Ακολουθεί τώρα η 202 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 του εισηγητού υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται και αυτή. 206 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Ο πρόεδρος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε παρήθευση. 207 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πάλι μια παραπάνω κάρτα για το Λαϊκό Κόμμα. Πέρας. 36 υπέρ, 29 κατά. Έχετε δίκιο κύριε Σουλίτερ. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210. Ε, συγγνώμη, απορρίφθηκε αυτή η 211. 210 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, επαλήθευση, επαλήθευση ηλεκτρονική για την 216 ψηφίσατε πέρας πάλι μία παραπάνω του Λαϊκού Κόμματος Φροντίστε παρακαλώ, γιατί πρέπει να ξαναγίνει τώρα η επαλήθευση. Αρχίζει πάλι λοιπόν η ψηφοφορία. Έχει ανοίξει πάλι η ψηφοφορία. Τροπολογία 216. 216. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Όχι. Ακόμη όχι. Ακόμη λείπουν πέντε. Τώρα κλείνει. 31 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. 219 του ισχύδου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται αυτή. 220 και 22 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το παράδειγμα τώρα 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 Α, έπρεπε και τις δύο να ψηφίσουμε μαζί. 62 και 2.38 είναι σχεδόν ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 2.39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στις αιτιολογικές σκέψεις. Ε, πρώτα ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχει καλυφθεί τώρα 68, 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά, εποχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται και αυτή. 73 Α, με συγχωρείτε, Πρώτα, η συμβαστική 13. Πρώτα βεβαίω, Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα η 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Α, ας, ας την επαναλάβουμε, ας την επαναλάβουμε. 78 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, βεβαίως η πλειοψηφία είναι υπέρ της απορρίψεως. Ενοποιημένη 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία που όπως πάντα γίνεται ονομαστικά, δηλαδή με ηλεκτρονική κάρτα, αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πάλι μία κάρτα παραπάνω από τον αριθμό των μελών του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή να βγάλει ε, κάποιος την κάρτα του. Τώρα έλεξε η ψηφοφορία. 55 υπέρ, 10 κατά και καμία άποχη. Συγχαρητήρια κύριε Παλέτσκης. Wir kommen jetzt zum Punkt 8. 8. Τώρα το θέμα 8. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την επόμενη έκθεση. Πρέπει να έχουμε μια αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω στις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, έτσι. Να μας εξηγήσει παρακαλώ ο εισηγητής. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Στο ΕΛΚΑ όντω υπάρχουν κάποιες αλλαγές στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ψηφίστε σύμφωνα με τις δικές μου οδηγίε παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα και αρχίζουμε με την τροπολογία 46. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαγμένη τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 54. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 30 υπέρ, 36 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. απόχέ, συγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά και για την 65 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Έλκα, άλλη μια φορά, άλλη μια φορά βλέπω ότι ψηφίζει ένας παραπάνω από σας. Φτάνει πια, λέει ο πρόεδρος. Πάντα έχουμε ένα παραπάνω. 40 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε για την 66 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τις ψηφοφορίες. 32 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Με 6 αποχές. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμός 7. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε θέλετε για την 80, ωραία. Ελέγχουμε για την 81 παρακαλώ, ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορία. 39-27. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε 90. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία. Ψηφίσατε όλοι. 90, έτσι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 33 υπέρ, 31 κατά εγκρίνεται. 91 υπέρ. 91 κατά εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται με μικρή πλουσία. 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Επαληθεύουμε λοιπόν για την 116. Ε, Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 32 υπέρ, 35 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας. Εντάξει, η γραμματεία θα φροντίσει. 35-32 έλεγα ότι ήταν το αποτέλεσμα. 35 κατά δηλαδή, οπότε απορρίπτεται. Συμβιβαστική αριθμός 11 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Η συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μικρή πλειοψηφία. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την 136 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 17 ψήφοι υπέρ, 49 ψηφί κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε για την 139. Ωραία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 139 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 34 ψήφοι υπέρ, 32 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η 139, 140 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε για την 140, εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της υποφορία. «33 ψήφοι υπέρ και 33 ψήφοι κατά και μία αποχή». Απορρίπτεται λοιπόν. 33-33 είναι το αποτέλεσμα. 141 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 143. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 34 υπέρ, 32 κατά. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145. Εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές. Ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155. Α, θέλετε να παληθεύσουμε. Ωραία. 154. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. 154. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίφθηκε. 21 ψήφοι υπέρ, 34 κατά και 3 αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161. Εκπίπτει. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 166. Θέλετε να επαληθεύσουμε για την 165. Καλώς. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41 ψήφοι υπέρ, 26 κατά. Καμία αποχή. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα από το ζητώ συγγνώμη. Η 165 εγκρίνεται λοιπόν. 166 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Στις αναφορικές σκέψεις. Κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε για το 6α. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα παληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 33 ψήφοι υπέρ, 31 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, ε, αποχές ελέγχουμε για την τροπολογία ρυθμός 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας.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 κατά, αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμός 13 παρακαλώ. Ψηφίστε. Δεν φαίνεται από εδώ καθαρά το αποτέλεσμα. Πέρα στις φοφορίες. 49 κατά 16 υπέρ. Καλά, καλά. Ε, σηκώνετε τότε τα χέρια σας καλύτερα για να μπορώ να σας βλέπω από εδώ. Συνεπώς απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. 14 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Αλλά θέλετε να επαληθεύσουμε γιατί 14. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά 14. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 33 κατά, 2 αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 15 παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 32 κατά. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε για την 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ισοψηφία 33-33. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Οι δύο τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν πενήντα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 24. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορία. Απορρίπτεται. 31 ψήφοι υπέρ, 34 κατά, μία αποχή. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, «26. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ γιατί δεν είναι σαφές από εδώ. Πέρας τις ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 50 κατά. Μία αποχή. Ειλικρινά, συναδελφοί, κάντε την προσπάθεια να σηκώνετε τα χέρια σας για να αποφεύγουμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και να χάνουμε έτσι χρόνο. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Και έτσι τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε για το τροποποιημένο σχέδιο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Με 63 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και μία αποχή. 63 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Σιγητά. Τώρα ψηφίζουμε την, ε, το σημείο 17. Κένεμπαχ. Έκθεση της κυρίας Κάντενμπαχ. Αρχίζουμε ευθύ αμέσως, για να μην χάσουμε και χρόνο, στην ψηφοφορία. με τις τροπολογίες 97, 98, 104, 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τρο... Παρακαλώ λέει ο πρόεδρος, με το σφυράκι δηλαδή. Τροπολογία υπαρθμών 100 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. πέρας υπέρ 32 κατά 19 101 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 της ίδιας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 12 της ηγετρίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεν είναι σαφέ, όμως. Ψηφίζεται Ονομαστικά, ηλεκτρονικά δηλαδή. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Υπέρ 34 κατά 24 εγκρίνεται. 115. 116 τώρα υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. 116. Ψηφίσατε. Πέρας. Απερίφθη με σημαντική πλειοψηφία. 20 προς 37. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ του εισηγητού. Ε. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά Πέντε συνάδελφοι συμμετέσχουν στην ψηφοφορία. Να ξαναψηφίσουμε τη 15 τι λέτε. Υπέρ λοιπόν, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές όμως, επαλήθευση. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρασε. 28 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Το δείχνει και ο πίνακας, εντάξει. 122 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 20 έχει αποσυρθεί. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Αυτή εκπίπτει. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά ηλεκτρονική παλήτευση, παρακαλώ αρχίζει ψηφίσατε Τέλος. Υπέρ 33 κατά 23. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Καλά. Επαλήθευση για την 25. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Την 25. Ηλεκτρονικά μου λείπουν τέσσερις συνάδελφοι αν θέλουν να συμμετάσχουν. Πέρας. 32 υπέρ. 26 κατά. Και καμία αποχή. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονική επαλήθευση. 133 αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. 46 υπέρ, 11 κατά. Άρα εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση πάλι 27 ψηφίσατε «44 υπέρ, 13 κατά». Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια. 28 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Καλά. 30 λοιπόν. Ψηφίσατε. Πέρασε. 50 51 ψήφοι. Πέρα 7 κατά. Και καμία αποχή. Είναι πιο δραστήριοι αυτοί που λένε όχι. Σηκώνεται λοιπόν καλά τα χέρια. Έχει πάντως Εγκριθεί σαφώ. 137 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Αλλά ας επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε. 137 λοιπόν ηλεκτρονικά. Πέρας. 34 υπέρ, 25 κατά, άρα εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 34 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται η 36. Τώρα, 37 με προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί 140, 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Α, θα επαληθεύσουμε την 38. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 33 ψήφι υπέρ, 24 κατά. Και μία αποχή. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 και 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 100... 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 και 148 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 149 υπέρ, κατά, αποχές. Ας υπαλληθεύσουμε γιατί είναι λίγο ασαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε, 149 λοιπόν ηλεκτρονικά, τέλος. 31 ψήφοι υπέρ και 29 κατά εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. 46 λοιπόν. 46 ηλεκτρονικά. Πέρας. 27 υπέρ, 32 κατά, απερίφθη 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Θέλετε επαλήθευση της 151. Καλά λοιπόν. Και πάντως παρακαλείστε όλοι να σηκώνετε καθαρά τα χέρια. Ψηφίσατε όλοι. Μου λείπουν ένα ή δυο ακόμα. Τέλος. 32 υπέρ, 28 κατά. Έγκρινεται. 47 εισηγείται υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 σε δύο μέρη, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 159 και 162 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 160 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 καλά. Επαλήθευση για την 164, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Πέρασε. Σαφέστατο το θετικό αποτέλεσμα, 40 υπέρ 19 κατά και μια αποχή. Η... Αγαπητέ Ζέμπερ, αυτοί που λέτε όχι, είσαστε πιο δραστήριοι, αυτό το ξαναλέω. 165 υπέρ, κατά. Επαλήθευση και εδώ, 165, γιατί δεν βλέπω καθαρά το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε, πέρασε. 28 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. 166 σε δύο τμήματα. Εγώ έχω το λόγο, έτσι είναι. 166 λοιπόν, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 167. Εκπίπτει έτσι είναι. 168, 69 και 70, όλες μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 171 έχει αποσυρθεί, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 100 Θέλετε επαλήθευση. 172. Επαληθεύουμε. Ψηφίσατε. Πέρας. 21 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175. Μόνο το δεύτερο τμήμα, ε, 175 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Ζητήθηκε επαλήθευση. Ναι, καλά. 176 λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 31 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 100 Νομίζουμε ότι κάποιος λέει τσεκ. Καλά. 56 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 28 υπέρ, 28 κατά. Απερίφη. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 ε, υπέρ. Α, 185, κάποιος ζήτησε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, αρχίζει, ψηφίζετε, ψηφίσατε όλοι. Μου λείπουν τρεις συνάδελφοι, δύο. Πέρασε. 27 μάλλον υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές. Καλά. Λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία για την επαλήθευση. Ψηφίσετε. Πέρας. 36 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίθηκε. Η 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 60 έχει αποσυρθεί, η 190 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και η 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 192 σαν του χάσει υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρο. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. 17 μόνον υπέρ, 44 κατά. Απορρίπτεται σαφέστατα. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε όλες μαζί 966 όλη αυτή τη λίστα που βλέπετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 100 209 μάλλον. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 212 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 72 και 214 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται. 213 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.15. Θέλετε επαλήθευση. Καλά, 213. Ψηφίσατε. 213, ονομαστική. Οι σοσιαλδημοκράτες, μία κάρτα παραπάνω. Καλά λοιπόν. Πέρας. 38 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ας κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για επαλήθευση. Ψηφίσατε. Πέρας. 25 υπέρ, 32 κατά, απερίφθη. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 226 λοιπόν ηλεκτρονικά ψηφίσατε. Πέρασε. 13 υπέρ 46 κατά. Οι κόκκινοι έχουν την πλειοψηφία. α το πω έτσι. 75 υπέρ. Κατά. Οποχές. Δεν είναι σαφές. Δεν είναι σαφές. 75 λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Πέρας. 31 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας η αιτιολογική σκέψη 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μαζί με την 84. 83 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές επαλήθευση της 83 ψηφίσατε την 83 ηλεκτρονικά πέρας 33 υπέρ και 26 κατά 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Α, εκπίπτει. Ερχόμαστε λοιπόν στην ψηφοφορία του συνόλου της γνωμοδοτήσεως που γίνεται ονομαστικά βέβαια. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 30 υπέρ, 11 κατά και 18 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότηση. Και συγχαρητήρια στην κυρία Κάντενμπαχ για την εργασία της. Έκθεση Γιώργενσεν. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκπίπτουν ορισμένες και ερχόμαστε στην τροπολογία 89 σαν του χάσει υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ενοποιημένη 2, ψηφίσατε, Φέρας. Φέρας είπα. 34 υπέρ, 25 κατά. 21 υπέρ. Κατά. Ε, υπέρ, ε, αποχές έγκρινεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. 9, ε, πρώτα την 22 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 37 κατά απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάλι τρία δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκπίπτουν πάλι ένας αριθμός από τροπολογίες και πηγαίνουμε στις 108 της κυρίας Μάνερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Πηγαίνουμε στην 6 υπέρ. Πρώτο τμήμα της 6. Κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 2 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τώρα προχωρούμε στην 7 ενοποιημένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και συνεχίζουμε με την 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε 36, 42, 43, 61, όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Απερίφθη λοιπόν το σύνολο αυτό. 44 υπέρ. Α, 150, μάλιστα. 150 ψήφι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, 37 υπέρ, 24 κατά. Καλά που κάναμε την επαλήθευση, εγκρίνεται. 151, 53 και 54 όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. 28 υπέρ, 31 κατά και μία αποχή. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Τροπολογία 1 δηλαδή. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, θέλετε επαλήθευση, καλώς 58 επαλήθευση ψηφίσατε πέρασε απερίφθη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 8, 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Επαλήθευση. Επαλήθευση για την 59. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ 30 κατά. Και μια αποχή. Απερίφθη. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Α, εκπίπτει, εκπίπτει. Καλά. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Πέρας. 33 υπέρ, 16 κατά και 12 άποχες. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια αγαπητέ κύριε Γιώργενσεν. Προχωρούμε αφού μας αρέσει τόσο πολύ η δημοσιονομική προοπτική. Η κυρία Ματίας είναι η συγγετρία. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Τσεκ λέει κάποιος. 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 29 έναντι 28. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 σε 2 τμήματα. Α, ηλεκτρονική επαλήθευση για το, την πέμπτη τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 6 κατά εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Μάλιστα. 6 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά του 8 ψηφίσατε όλοι ένας παραπανήσιος έχουμε στους σοσιαλιστές Εγκρίνεται 29 υπέρ. 9. Ποιοι είναι υπέρ. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας 34 υπέρ, 21 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, υπέρ κατά αποχές 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 έχει καταπέσει και 18 έχει καταπέσει. 22 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 22. Τέλος της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 19 δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ. Ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συγκεντρωτική 1. Τι θέλετε να επαναληφθήσουμε την 25. Μάλιστα ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 27 υπέρ 26 κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, συγκεντρωτική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. ist abgelehnt. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε τη 38. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, η συγκεντρική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, Α, να επαληθεύσουμε. Ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος στη 43. Ψηφίσατε όλοι. 32 υπέρ, 27 κατά, εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός για τις 45. Ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι.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 Τέλος ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 45 κατά. Και μία αποχή. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, με συγχωρείτε. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 και 63 Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61 ζητήθηκε. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. 61. Για την 61 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 30 υπέρ 24 κατά 6 εποχές εγκρίνεται. 62 και 63 μα από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 έχει καταπέσει, 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στην εισηγήτρια. 56 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, μια αποχή. Συνεχίζουμε, μιας που έχουμε πάρει φορά. Με την έκθεση Μακάβαν. Λίντα, θέλετε το λόγο. Όχι, απλά ένα διαδικαστικό έχω να κάνω, Πρόεδρε. Κανονικά υπέρ είναι πράσινο και κατά είναι κόκκινο το χρώμα. Κάπως μας μπερδεύει τώρα εδώ πέρα. Είναι ανάποδα τα χρώματα στις οθόνες. Ε, τι να σας πω, εγώ χαίρομαι που υπάρχει καν ο πίνακας και που λειτουργεί. Θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε βέβαια για το απόγευμα γιατί έχουν αλλάξει τα χρώματα. Ευχαριστώ πάντως για την επισήμανσή σου. Ερχόμαστε στην απαλλαγή για την ΕΦΣΑ, τροπολογία 1, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, Δεύτερο. Ε, μάλλον κατά αποχές. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 έχει αποσυρθεί, 7 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 8 υπέρ,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 αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική Ψηφίσατε. Πέρασε. 44 υπέρ, 4 κατά και 8 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η απαλλαγή για την ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια κυρία Χάουκ. Συνεχίζουμε αμέσως. Και προχωράμε στην ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Φάρμακα. Απολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πέντε. με μια τροπολογία προφορική Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 7 έχει ε, αποσυρθεί, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, το 10 έχει αποσυρθεί, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 48 ψηφί υπέρ 7 κατά μία αποχή. Και έχουμε εδώ πάλι πολύ ενδιαφέροντα ε, χρώματα που εμφανίστηκαν στην οθόνη.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 49 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Μπράβο κυρία Χάουκ. Τέλος της ψηφοφορίας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την πειθαρχία τους. Και επειδή περάσαμε τόσο ωραία θα το διασκεδάσουμε και στις 3 με συνέχεια των ψηφοφοριών. Γεια σας και καλή όρεξη.